Der Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Präsident war pünktlich und deswegen habe ich gesagt... Καλώς ήρθατε. Ας αρχίσουμε, έστω και αν δεν είναι παρόντες όλοι οι αρμόδιοι. Βλέπω ωστόσο τον Επίτροπο Ζακ Μπαρό και του απευθύνω το καλώς ορίσατε. Ελπίζω και η Προεδρία του Συμβουλίου να προσέλθει. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση λοιπόν. Το πρακτικό της χρησινής συνεδριάσεως έχει ήδη διανεμηθεί. Ερωτώ εάν έχετε ενστάσεις. Όχι. Καλώς λοιπόν εγκρίνεται το πρακτικό. Ακολουθούν δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών για την επανεισδοχή πρώην κρατουμένων του Γουαντάναμου. Εξ ονόματος πρώτα βέβαια της Προεδρίας λαμβάνει το λόγο ο Υπουργός κ. Φόρντρα. So,